17 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προέβη σύμφωνα με τον κανονισμό Ανακοινώσει είναι λοιπόν διάρκεια τη συνεδρίαση τη 12η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προέβη, σύμφωνα με τον κανονισμό, στην εξέταση συμβατότητας της πράξης, της, με την πράξη της 20 Σεπτεμβρίου 1976 της προσωρινής αποστολής που αν, ανέθεσε ο Γάλλος Πρωθυπουργό στον κύριο Αγνόν Ντανζόν αναφορικά με την έναρξη εκπόνησης μιας στρατηγικής αναθεώρησης εθνικής άμυνας και ασφάλειας και αποφάσισε τελικά η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ότι η αποστολή αυτή